έχω μια ανακοίνωση να σας κάνω. Από την GUE έχω λάβει αιτήματα για διορισμούς σε επιτροπές και αντιπροσωπείες. Ο κατάλογος θα επισυναυθεί στα πρακτικά. Και αν δεν υπάρξει αντίρρηση κατά την έγκριση θα